Uh, good morning everybody. I will now start the meet. Καλημέρα, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Change to Swedish before we go to the... Και θα μιλήσω μετά σου ειδικά πριν ξεκινήσουμε τη συμφορία. Hej och välkomna allihopa. Ni är jättevälkomna. Καλώς ορίσατε όλοι στη σημερινή συνεδρίαση και το πρώτο σημείο είναι η έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, δεν έχουν κατατεθεί προτάσεις ε, τροποποίησης του σχεδίου ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Το σημείο 2 τώρα είναι οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή ότι στις 12 Νοεμβρίου αυτή η μισή ημέρα που έχουμε ακυρώθηκε, δυστυχώς. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και δεν έχουμε αρκετό χρόνο, ε, αλλά δεν υπάρχει θέση. Τι να κάνουμε. Δεν έχω άλλη ανακοίνωση και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις συστάσεις ε, των συντονιστών. Έχουμε τα πρακτικά από τις συνεδρίες των συντονιστών στις 19 Σεπτεμβρίου. δεν υπάρχουν ενστάσεις θεωρούνται εγκεκριμένα. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 4. Θα ήθελα παρακαλώ να μην κάνετε τόση βασαρία ή δυνατόν για να αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία παθήσεων των γυναικών. Η κυρία Αγγελίλη, η θα ήθελε ίσως να πάρει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρα από το ότι θέλω προφανώς να ευχαριστήσω όλες τις συναδέλφους για τη μεγάλη επικοδομητική συμμετοχή τους σε εργασίες, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση πάνω απ' όλα που αφορά την τροπολογία 33 που εγώ ίδια υπέβαλα εξάλλου. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα μεταφραστικό σίγουρα στην αγγλική μετάφραση. Στο κείμενο στα Ιταλικά γράφεται η υγειονομική βοήθεια, πρωτοβάθμια βοήθεια, υγειονομική βοήθεια. Στη μετά στην αγγλική λέει ιδιωτική περίθαλψη. Δηλαδή πρωτοβάθμια μεταφράστηκε σαν ιδιωτική. Ε, προφανώς λοιπόν δεν είναι σωστή μετάφραση. Ε, γνωρίζω ότι θα γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Θα ήθελα να γίνει έλεγχος των μεταφράσεων ε, διότι μιλάμε για πρωτοβάθμια ε, βοήθεια που παρέχεται περίθαλψη και όχι ιδιωτική περίθαλψη. Ευχαριστώ πολύ, Λεπρόεδρος. Είναι πολύ καλό που το διευκρινίζετε διότι πρόκειται περί πραγματικά διαφορετικών ενιών. Private και primary. Ε, και εγώ όπως το βλέπω είναι διαφορετικό. Ε, ρωτώ, οι πράσινοι εξακολουθούν να θέλουν ψηφορία κατά τμήματα, το split vote. Οι πράσινοι το ζήτησαν. Το θέλετε. Έτσι, δεν λέμε private, αλλά primary εδώ, ε, στο αγγλικό κείμενο. Οπότε, εντάξει, το αποσύρεται, έτσι. Εντάξει, καλώς. Οπότε, δεν θα γίνει στην τροπολογία 33 ψηφοφορία κατά τμήματα. Okay, we don't start to vote and... Ωραία, να αρχίσουμε την ε, ψηφοφορία. Ε, τροπολογία 75, ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Ε, θα ξαναρχίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ με ανάταση κατά αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά αποχές, νομίζω ότι πρέπει να γίνει επαλήθευση για την τροπολογία 76, ε, του ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 77 με τμήμα, κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ,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 Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 89 υπέρ. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 και 94 είναι ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι 97 και 96 καταπίπτουν και περνάμε στην 99 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, οι 101 και 104 είναι ταυτόσιμες και έχουμε και κατά τμήματα ψηφοφορία. Θα αρχίσουμε με το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Δύσκολο να κρίνει κανείς την έκβαση. Θα κάνουμε παλήθευση για το δεύτερο τμήμα, γιατί σε 101 και 104. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Πέρασε. Είναι ξεκάθαρο ότι εγκρίνεται. 102. Θέλω να διευκρινίσω κάτι εδώ. Ε, στο δικό σας κατάλογο μπορεί να φαίνεται ότι πρόκειται για μία μόνο τροπολογία για 102 και μετά έχουμε κατατμήματα ψηφοφορία για την 103. Το αντίστροφο ισχύει. Η κατατμήματα ψηφοφορία είναι για την 102 και όχι για την 103. Αλλά είναι σωστό το κείμενο που αναγράφεται στον κατάλογο, αλλά πρέπει να το συνδέσετε με την 102. Με παρακολουθείτε, το καταλάβατε τι εννοώ, γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζετε. Θα κάνουμε κατά τμήματα ψηφοφορία για την 102 και όχι για την 103. Εντάξει. Πρώτο τμήμα για την 102 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 103 τώρα υπέρ, κατά, αποχές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 εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, αυτό σημαίνει ότι καταπίπτει μία σειρά τροπολογιών και φτάνουμε στην 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 και 123 είναι ταυτόσιμες υπέρ των δύο παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνονται. Αυτό σημαίνει ότι 122 κατά καταπίπτει. Ψηφίζουμε για την 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα μπορούμε να πάμε στην 134 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 καταπίπτει και ψηφίζουμε για την 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές ε, ε, εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω χρειάζεται επαλήθευση για την 153 ψηφίστε παρακαλώ για την 153 the vote is closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. 155 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Θέλετε παλήθευση για την 157. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed.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 κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, ψηφίζουμε για την 176 τώρα υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα... 185 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 καταπίπτει. 189 τώρα υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 189. The vote is closed. It's rejected. Απορρίπτεται. Uh, amendment 190. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα 22. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, κατεβαίνουμε στην τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Α, ξανά, παρακαλώ. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 33 Ε, δεν είναι πλέον κατά τμήματα η ψηφοφορία. Ε, φυσιολογική ψηφοφορία για την 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πρέπει να κάνουμε για την επαλήθευση. Δεν πρόλαβα να μετρήσω. 34. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. The vote is closed. Πέρας. Uh, okay. Is that really? <laughs> Okay, there has been something wrong with the translation because... Ε, είμαι πολύ γρήγορος και δεν με πρόλαβαν οι διερμηνείς μάλλον. Δεν πειράζει. Ε, ε, we then go to amendment... 36. Όχι 35, διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 και 38 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Yeah, so we have. We, we just go back. Yes, exactly. We have to go back to Δυστυχώς πρέπει να επιστρέψουμε στην τροπολογία 30. Την ξέχασα. Ήταν ανάμεσα στις τροπολογίες που κατέπεσαν. 30 ναι, παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. I 39 Στην 39 είμαστε, νομίζω. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές ένα λεπτάκι ξανά υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 πίπτη και ψηφίζουμε για την 56 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ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 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι καταπίπτει 67. Όχι, όχι, όχι δεν καταπίπτει. Τη ψηφίζουμε. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 τώρα υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται 70 υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται 72 υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση για την 72. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 72. Okay. The Εγκρίθηκε. Άρα καταπίπτει η 71 και περνάμε στην 73. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Γκρίνε. Μπορούμε ομού να ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες. Όχι, όχι. we take the rest of the in Ωραία, λοιπόν, για όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκαν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψηφίσουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is open, still open, and Περιμένουμε να ψηφίσουν και άλλοι. Δεν έχει κλείσει ψηφοφορία. Υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να ψηφίσουν. Ένας λείπει. Καλά, πέρασε. Σαφέστατα εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία μας. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία για την σεξουαλοποίηση των κοριτσιών. Η κυρία Κελέσκα, μήπως θέλετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις ε, τροπολογίες που μας έστειλαν. Όπως ξέρετε, είχαμε 134 ε, τροπολογίες και ήμουν κατά 22 από αυτές. Όπως τα είδατε ήμουν αρκετά ανοιχτή ε, σε θέση να συνεργαστώ με όλες πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με τη διαγραφή της παραγράφου 11 όμως δυστυχώς δεν μπορώ να συμφωνήσω με την 76, την 92 και την 94 ε, που είναι τροπολογίες του Προέδρου και δεν τις υποστηρίζω διότι νομίζω ότι εξαετή και ετή κορίτσια δεν είναι έτοιμα να διδαχθούν για την αναπαραγωγική υγεία, για τα δικαιώματα αναπαραγωγής και για την αντισύλληψη. Όμως για όλες τις άλλες τροπολογίες σας ευχαριστώ και ελπίζω να υποστηρίξετε την έκθεσή μου. Okay, we will Καλώς, θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θέλω να πω ότι η συγγήτρια θεωρεί ότι υπάρχουν λάθη στον κατάλογο ψηφοφοριών Θέλετε να το διευκρινίσετε το θέμα όταν φτάσουμε στην τροπολογία 94 ότι έπρεπε να είναι μάλλον ε, προστίκη η 94. Περί αυτού πρόκειται. Ναι. Θα σας δώσουμε το λόγο όταν ε, θα θέλετε να το διευκρινίσετε. Ξεκινάμε με την τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές πρέπει να ελέγξουμε την 45 άρχεται η ψηφοφορία ο έλεγχος ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο έχουμε Πέρα ψηφοφορίας δεν ξέρω ίσως πρέπει να επαναλάβουν την ψηφοφορία, διότι έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ περίπου παραπάνω. Αχα, Okay. Okay. Καλώς. You can put in we take vote again. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις 45 την τροπολογία 45. Ξεκινάμε. Ελάτε, ελάτε. Τέλος ηχοφορίας. Εγκρίνατε. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 Αποσύρεται. 49 δεν ψηφίζουμε. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Εκτός μικροφώνου κάτι ακούγεται. Εμείς δεν ακούμε. Οι Δεν είχα χρόνο να τη δω. Έφτασε αργά χθες το βράδυ. Έχω αντίρρηση λοιπόν. Υπάρχει μια αντίρρηση ότι αυτή η περιπτώση δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Πάμε στην τροπολογία 48 υπέρ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα η προφορική, οι τροπολογίες 57 και 52 καταπίπτουν. Πάμε στην... Αποσύρεται η 56, 55 και 58 δεν ψηφίζουμε. Πάμε στην τροπολογία 59. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπορεί να γίνει έλεγχος βεβαίως, ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 59. Ξεκινάει η ψηφοφορία. The vote is closed. It's rejected. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 63 και έχουμε προφορική τροπολογία Υπάρχει αντίρρηση κατά τη προφορικής τροπολογίας. Θα ήθελα να προβάλλω αντίρρηση εκ νέου διότι δεν την έχω δει. Καλώ, ο Πρόεδρος, οπότε προφορική τροπολογία καταπίπτει και πάμε στην τροπολογία 64. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, έλεγχος για την 65. Ξεκινά ηλεκτρονικό έλεγχο για την 65. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 καταπίπτει και 66 ψηφίζουμε την 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Έλεγχος για την 69 βεβαίως. Ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 69. Πέρας. Εγκρίνεται. 71 ε, in... Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 71 έλεγχος. Ξεκινάει. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ίσως θα είναι εύκολο να ελέγχουμε συνέχεια. Πιο εύκολο. Δοκιμάζουμε έτσι και βλέπουμε. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 72. Ίσως να είναι ίδιο το αποτέλεσμα. And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να έχει απορριφθεί, ε. δεν βλέπετε, δεν σηκώνετε το χέρι σας. Έλεγχος για την 73. Ξεκινάει. Πέρας. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Ελέγξαμε τις περισσότερες. 74 έλεγχος ηλεκτρονικό, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα κάνουμε αυτό κατευθείαν ηλεκτρονική ψηφοφορία. 74. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα οι 76, 81, 75, οι 82 καταπίπτουν και πάμε στην τροπολογία 80. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 80. The vote is closed. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 83 Κάνουμε έλεγχο κατευθείαν η τροπολογία 83, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η κυρία Γιανακουδάκη απερίφθη, η τροπολογία της κυρίας Γιανακουδάκη μάλλον, απερίφθη. Ψηφίζουμε την τροπολογία 84, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 84. Ξεκινάμε στην 84. Mm, okay. The vote Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, that means a lot of... Ε, we can go down amendment 90. Πάμε στην 91 τώρα. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την τροπολογία 91 The vote closed. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 92 Με δύο ψήφους διαφορά υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 94. Προφορική τροπολογία. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, στην εισηγήτρια που θέλει να κάνει κάποια διευκρίνηση, θέλει να κάνει κάποια προστίκη. Εισηγήτρια. Όχι, όχι, λέει η εισηγήτρια. Όχι, πραγματικά, δίκιο έχετε, τα πάντα είναι εντάξει στον κατάλογο ψηφοφοριών, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί αυτή την περίπτωση, λέει ο Πρόεδρος, ε, λέω υπάρχει αντίρρηση κατά των προφορικών αυτοτροπολογίων, τη προφορικής τροπολογίας. Όχι. Okay. Ε, do you want to ξεκαθαρίσετε ποια είναι περί τίνος πρόκειται αυτή η προφορική τροπολογία. vote. It's just split vote, yeah. So it's an it's a, it's an yeah, but it's an addition to yeah. If you look in the, in, in the last... Αν δείτε στην τελευταία σελίδα του καταλόγου ψηφοφοριών, η συγγήτρια. Κυρίες και κύριοι, στο τέλος του καταλόγου, παράγραφο 10, λέμε αυτό που ενδείκνεται στην ηλικία, appropriate to age, το ενδεικνυόμενο για την ηλικία. Σεξουαλοποίηση που είναι η ενδεικνυόμενη για την ηλικία, που αντιστοιχεί στην ηλικία. Δεν θα ψηφίσουμε προφορική τροπολογία, λέει ο Πρόεδρος. Θα έχουμε στον κατάλογο ψηφοφορία την προφορική τροπολογία αυτή καθ' αυτή. Αργότερα στην τροπολογία 95 έχουμε την προφορική τροπολογία. Σωστά τα είχαμε εξ αρχής στην, κατάλογο. Δεν έχουμε στην 94 την προφορική τροπολογία, αλλά μόνο κατά τμήματα στην 94 τώρα ψηφίζουμε. Εντάξει, με καταλαβαίνετε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 94 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ίσως να ήμουν πολύ γρήγορος. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Έλεγχος λοιπόν. Για το δεύτερο τμήμα ξεκινάει ηλεκτρονικός έλεγχος. The vote is closed εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 αποσύρεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά έχουμε προφορική τροπολογία της κυρίας Κρυλεύσκα υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά την προφορική τροπολογία Έχετε αντίρρηση. Εν τη αυτή περίπτωση δεν θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Προχωρούμε. Πάμε στην τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 98. Ξεκινάμε τον ηλεκτρονικό έλεγχο για την 98. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα καταπίπτουν πολλές τροπολογίες και πάμε στην τροπολογία 104 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε την 104. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 104, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 11 λέει εδώ. Κατά τμήματα, ξεχωριστά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107 υπέρ. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Προχωράμε και πάμε στην 110 λοιπόν. 110 υπέρ κατά άποχες νομίζω ότι εγκρίνεται έλεγχος για την 110 ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 110 τέλος απορρίπτεται ζητώ συγγνώμη γι' αυτό συμβαστική 3 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται άρα πάμε στην 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 115 ξεκινά για την 115 τέλος εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι χρειαζόμαστε έλεγχο για την 131 ξεκινάει ηλεκτρονικός έλεγχος τέλος απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται έλεγχος για την 134 ξεκινάει τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 και 5 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε την 7 ξεκινάει ηλεκτρονικός έλεγχος η τροπολογία 7 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 Α, ναι, δίκιο έχετε. Ναι. Καταπίπτει. Πάμε στην τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 14 έλεγχος για τη 14 ξεκινάει η ψηφοφορία τροπολογία 14 ηλεκτρονικός έλεγχος τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται αλλά ήταν πραγματικά μηδαμινή διαφορά τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 δεν ψηφίζουμε ψηφίζουμε 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Έλεγχος λοιπόν για την 20. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 20. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Βλέπω τον αριθμό των χεριών μόνο. Δεν κοιτάω τους συντονιστές, δεν κοιτάω τίποτα άλλο διότι λένε ότι πρέπει να κοιτάτε τους συντονιστές, αλλά δεν αληθεύει. Κοιτάω εσάς, αν δεν σηκώνετε τα χέρια και δεν το δω με τα μάτια μου τα ίδια, αν δεν βλέπω τα χέρια σας, αν δεν τα σηκώνετε δεν τα βλέπω. Είναι απλούστατο. Χαίρομαι που ελέγχετε, είναι πολύ καλό. Αν είστε αβέβαιες, εντάξει, ζητάτε να γίνει έλεγχος. Ή θα το ξεκαθαρίσω αυτό. Πάμε στην τροπολογία 22. 22 υπέρ κατά αποχές σαφώς εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 23. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 23. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 26 υπέρ. Κατά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 για την 36. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 36. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 37. Ξεκινά ο ηλεκτρονικός έλεγχος για την 37. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 38. Από την αρχή ηλεκτρονική ψηφοφορία για 38. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. 38. Τέλος. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 39 αποσύρεται. Πάμε στην τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα τα κάνουμε έλεγχο έλεγχος λοιπόν γιατί 42 ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφόρια τέλος απορρίπτεται με τέσσερις ψήφους διαφορά wow τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του και ξεκινά η ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος. Τέλος ψηφοφορίας. Και το ψήφισμα απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 14-12. Πάμε στο επόμενο σημείο, 6 ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2011 και την πολιτική τη σχετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πολιτική όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία. Η κυρία Γκάμπριελ θέλει να πάρει το λόγο. Ξεκινάμε την ψηφοφορία και ξεκινάμε από τη συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδικά. Ψηφίζουμε τη 19 τώρα. Ποιος είναι υπέρ της 19. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την τροπολογία 1. Ξεκινά η ψηφοφορία για την 1. The vote is closed. Πέρασε, απορρίπτεται. Then I ask, can we take the rest of in block? Λοιπόν, τις υπόλοιπες τροπολογίες μαζί, να ψηφίσουμε. Όλες εκτός από την 8, μαζί. Όλες μαζί εκτός από την 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα. Όλο στο σύνολό του. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Σαφώς εγκρίνεται. Μετά. Έχουμε κατάλληλη ψηφορία για πρόγραμμα κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την περίοδο 2014 μέχρι 2020 το πρόγραμμα δικαιοσύνη. Λοιπόν, πρόγραμμα δικαιοσύνη για την περίοδο 2014-2020. Η συγγήτρια θέλει να πει κάτι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τι ψηφοφορίε. Τροπολογία 4. Μετά την τροπολογία 26 μπορούμε να τις εξετάσουμε όλες μαζί, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Πέντε 28 Από την 28 και πέρα, λέει ο Πρόεδρος. Μαζί.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 Πάμε στην τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τροπολογία 7. Ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα 25-26 καταπίπτουν. Πάμε στην 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. No okay. 28. Uh, uh, Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για τη 33 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται Τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του ξεκινάει η ψηφοφορία Πέρα ψηφοφορίας και σαφώς εγκρίνεται και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια μετά πάμε στην 8 ειδικό πρόγραμμα εφαρμόζει τον ορίζοντα 2020, Horizon 2020. Uh, Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απόχειας. Ε, ξεκάθαρα εγκρίνεται. And then we have the, the nine proposal for regulation on European statistic on demography. Τώρα περνάμε στην πρόταση κανονισμού για τις νέα στατιστικά στοιχεία, για ε, νέα στατιστικά δημογραφικά στοιχεία. Όλα μαζί παρακαλώ υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Good luck.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 I will now start... Θα συνεχίσουμε τώρα τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ, καθίστε. If you please take your seat and if you... παρακαλώ. I will now change over to Swedish. Και θα αρχίσω να μιλάω και σουηδικά. You really think you need to talk? You can do it outside. Ε, αν θέλετε ντε και καλά να μιλήσετε, έχει μπόλικο χώρο απ' έξω, ε, πηγαίνετε έξω να μιλήσετε. Okay. Θα μιλήσω σου ειδικά όπως θα καταλάβατε ήδη. Έχουμε μια επίσκεψη από ένα κλιμάκιο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Πρόκειται για μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Οικογένειας Ηλικιωμένων Πολιτών, Γυναικών και Νέων της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ε, προσβλέπουμε συζήτηση, θέλουμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Η κυρία Βέλκιν Φάρ, Κρίστελ Φούρνεν, Μόνικα Λασάρ, και η κυρία Συμπιλάουρης φυσικά που είναι η πρόεδρος ε, της Εν Λόγω Επιτροπής είναι σήμερα μαζί μας ε, και στις 3 ε, Οκτωβρίου ήσασταν και εσείς εξάλλου στη μεγάλη μας διάσκεψη. Σας καλωσορίζομαι και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συσφίξουμε τους θεσμούς ανάμεσα στους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς βουλευτές. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ουσιαστική ανταλλαγή απόψε. Είναι τέλειο που ήρθατε σήμερα και θα... Θα δώσω το λόγο πρώτα στην Πρόεδρο, να κάνετε την πρώτη σας παρέμβαση και μετά θα αφήσουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να λάβουμε θέση εδώ σύντομα. Ως αντιπροσωπεία της Επιτροπής Οικογένειας ηλικιωμένων γυναικών και Νεολαίας της Γερμανικής Βουλής Έχουμε έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενημερωνόμαστε για θέματα πολιτικής ισότητας των φύλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας και επανειλημμένα το έχει τονίσει άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε όλη την Ευρώπη χρειάζεται ποσόστοση για τη συμμετοχή των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Εμείς το επιθυμούμε. Στη Γερμανική Βουλή το θέμα αυτό είναι αφιλεγόμενο Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει όλους ιδιαιτέρως να ακούσουμε πώς έχει η συζήτηση και οι θέσεις για το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς προχωράει αυτή η ε, συζήτηση. Αντίστοιχε συνομιλίε είχαμε χτε με την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ αλλά και με βουλευτές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ένα άλλο θέμα ε, που μας ενδιαφέρει από πολιτικής ισότητας γυναικών είναι κατά την άποψή μας επίσης πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της μισολογικής ψαλίδας ε, με βάση το φύλλο. Και αυτό Υποστηρίζεται ε, σε κοινοτικό επίπεδο από αντίστοιχη οδηγία. Στη Γερμανία έχουμε ακόμα να κάνουμε κάποια δουλειά γιατί δεν αμοιβώνται το ίδιο άνδρες και γυναίκες ενώ κάνουν την ίδια εργασία. Αυτό είναι ένα έλλειμμα και δείχνει ε, τι σημαίνει ισότητα των φύλων και πόση δουλειά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Και οι λύσεις είναι επίσης δύσκολο βρεθούν. Δεν το κρύβω ούτε το παραγνωρίζω αυτό. Βλέπω ότι η ανταλλαγή που έχουμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είναι σημαντική. Η διάσκεψη της 3ης Οκτωβρίου ήταν πολύ καλό μήνυμα και για μένα και κατά την άποψή μου είχε πάρα πολύ σαφείς στόχους θέση. Η ισότητα των φύλων είναι ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό ε, σήμα κατά τεθέν και πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ αυτή την εβδομάδα. Δεν συνεδριάζει τούτη τη εβδομάδα η Bundestag στο Βερολίνο. Γι' αυτό θα μπορέσουμε να μεταβούμε και στο Παρίσι και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις όχι μόνο στο Βέλιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και με τους Γάλλους γείτονές μας. Ε, είμαστε επίσης πρόθυμοι να σας δεχθούμε όποτε θέλετε να έρθετε στο Βερολίνο. Σταματώ εδώ και θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία να μιλήσουν και οι συνάδελφοί μου αν συμφωνείτε κι εσείς. Αλλά εσείς προεδρεύετε πρόεδρε, όχι εγώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να Α συμπληρώσω μόνο στα όσα είπε η κυρία Λάουρη στο εξή. Το θέμα των ποσοστώσεων των γυναικών σε ηγετικέ θέσει ε, και διοικητικέ είναι συμβολικό. Όσοι ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα ξέρουν ότι δεκαετίε περιμένουμε να κινηθεί λίγο η κατάσταση και δεν έχουν κινηθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό ο συμβολισμό. Και να ε, διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν και από τα κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να μπορέσουμε από κοινού να ε, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Χθε είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με την κυρία Ρέντεγκ και ελπίζω φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πρόταση αλλά θα είναι το πρώτο και μόνο βήμα αυτό και το θέμα είναι τι θα κάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις, τι θέση θα πάρουν σχετικά και βεβαίω τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να επηρεάσουν, ή μάλλον είναι ερώτηση αυτό, μπορούν να επηρεάσουν τη θέση της κυβέρνησης του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα για να προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι κάναμε τα τελευταία 40 χρόνια. επόμενη ομιλήτρια. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εγώ ε, για τις γυναίκες σε διευθυντικές σχέσεις. Για τις αμοιβέ δεν θέλω να πω τίποτα. Συμφωνούμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα ότι χρειάζεται περισσότερη δράση και στη Γερμανία αλλά και υποστήριξη από ευρωπαϊκής πλευράς. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα, ε, την οδηγία για την προστασία της μητέρας. Εχθές ε, και προχθές ακούσαμε ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί ε, έχουν ε, οδηγηθεί σε ένα διέξοδο αυτό τον καιρό. Και ε, μπορούσαμε ίσως να ακούσουμε από εσά και από την κυρία Εστρέλια από πρώτο χέρι τι δυνατότητες υπάρχουν ακόμα συμβιβασμού, διαπραγματεύσεων, γιατί είναι δύσκολο όταν κανείς δεν συμμετέχει άμεσα σε κάποιες διαδικασίες. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε της άμεσης επαφής μαζί σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε και τους βουλευτές που παρίστανται. Λούλινγκ. Η κυρία Λούλινγκ. Äh, <clears throat> ε, θα προσπαθήσω να το πω γερμανικά, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, σα από την Bundestag. Θα ήθελα σύντομα να απαντήσω στις σύντομες ερωτήσεις σας για τις ποσοστώσεις. Σε εμά το θέμα είναι εξίσου αμφιλεγόμενο και επίμαχο όπως και στην Bundestag και στο ιστορικό των πολιτικών ομάδων αλλά και μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ προβληματίζομαι και αναρωτιέμαι σε ό,τι αφορά το σύστημά μας, ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με ποσοστώσεις ε, στην πολιτική όταν το αποφασίζουν τα πολιτικά κόμματα αυτό. Ή όταν θεωρεί μια χώρα ότι θέλει να υπάρχουν ποσοστώσεις σε δημοσίους οργανισμούς. Αλλά δυσκολεύομαι λίγο και ε, ζορίζομαι με ποσοστώσεις στην ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Σε ιδιωτικές εταιρείες εμείς θα υπαγορεύουμε τι θα κάνουν. Υπάρχει και το εταιρικό δίκαιο που στην Ευρώπη διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εγώ είμαι από το Λουξεμβούργο. Δεν έχουμε και υποπτικά συμβούλια, έχουμε μόνο διοικητικά συμβούλια στις επιχειρήσεις. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό ως δομή. Και στα Προεδρία, έτσι κι αλλιώς στα Διοικητικά Συμβούλια και η κυρία Ρέντινγκ από το Λουξεμβούργο είναι. Και το συζήτησα. Γιατί εδώ στο Κοινοβούλιο τώρα το έχουμε κάνει ολόκληρη υπόθεση γιατί λέει να διοριστεί άνδρας στο Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και τη ρώτησα και μου λέει η κυρία Ρέντινγκ δεν πρόκειται να προτείνω για τέτοια προεδρία γυναίκες ποσοστώσεις. Δεν πρόκειται. Εδώ έχουμε την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή και θα γίνει ακρόαση κανονικά, γιατί από το Μάιο χειρεύει μία θέση ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Διευθυντικό Συμβούλιο, που είναι έξι. Ε, και από τους έξι η μία θέση χειρεύει από το Μάη. Ε, και όχι μόνο αυτό, εδώ και 1,5 χρόνο το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν υπάρχει γυναίκα. Και έχουν διοριστεί εκ τούτου τρεις άνδρες. Βέλγος, Γάλλος και Γερμανός. Ο αρνήθηκε την ακρόασή τους εδώ. Και μια χώρα που έχει 68 εκατομμύρια κατοίκους είναι πιο εύκολο να βρει μια γυναίκα από ότι μια χώρα με μισό εκατομμύριο, ε, από τους οποίους το 40% είναι και ροδαπή. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα, να είμαστε ισχυροί απέναντι στους αδυνάτους και δυνατοί απέναντι στους ανίσχυρους. Μάλλον ε, ε, και ανίσχυροι απέναντι στους δυνατούς. Και με αυτό το τσίρκο, πραγματικά έτσι θα το χαρακτηρίσω, που γίνεται γύρω από την υποψηφιότητα του κυρίου Μέρς, δεν κερδίζουμε τίποτα. Ούτε εξυπηρετούμε κανέναν στο κοινοβούλιο. Και μετά θα σου πούν, ρε, σου αφαιρώ και το δικαίωμα ακρόαση, κοινοβούλιο, θα έχεις μόνο δικαίωμα διαβούλευσης, να λες τη γνώμη σου και τελείωσε. Για θα αποφασίζει το Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δύναται. Και ξέρετε, εγώ είμαι η πιο ηλικιωμένη γυναίκα στο Κοινοβούλιο. Το 1965 ήμουν η νεαρότερη Ευρωβουλευτής και από τότε που πολιτεύομαι ασχολούμαι με γυναικεία θέματα, 40 και πλέον έτη τώρα. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε πετύχει διάφορα πράγματα, αλλά πάντα με τη λογική και όχι με παραλογισμούς τώρα, γιατί παραλογιζόμαστε πια σε διάφορους τομείς. Ναι, ναι, και στην προστασία των μητέρων. Ε, και με αυτό δεν πετυχαίνουμε τίποτα, πράγμα που αποδείχτηκε. Αυτά για τις ποσοστώσεις. Τώρα, για τη μισθολογική ψαλίδα, ε, με βάση το φύλλο, gender pay gap, όλα αυτά είναι μέση όρη και δεν έχει καμία αξία αυτό για την ίση αμοιβή, για ίση εργασία ή οτιδήποτε. Και στη χώρα μου υπάρχουν οδηγοί λεωφορείων, άνδρες, που κερδίζουν πολύ λιγότερα κερδίζουν πολύ λιγότερα χρήματα από άλλους άνδρες ε, οδηγούς λεωφορείων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες τους πληρώνουν λιγότερο, ενώ είναι άνδρες και οι δύο στη χώρα μου. Έγινε και μια στατιστική μεταξύ ε, για τις διαφορές πληρωμής αμοιβών των εργατών, έτσι, των χειρονακτών, ε, ανδρών και γυναικών στις διάφορες χώρες. Το Λουξεμβούργο είχε πατώσει. Για ποιο λόγο. Γιατί στη δική μας βιομηχανία κυριαρχούσαν η χαλιβουργία, και μάλιστα τα ορυχεία. Και οι γυναίκες που δούλευαν εκεί ήταν μόνο καθαρίστριες. Και βέβαια έβγαζαν λιγότερα από τον ε, υπερηδικευμένο ε, ανθρακορίχο ας πούμε ή ε, χαλιβουργό. Τι λέει η οδηγία. Η οδηγία είναι πάρα πολύ καλή. Θα μπορούσα να σας δώσω και παραδείγματα αλλά δεν ε, έχουμε χρόνο. Τι γίνεται ε, στο Λουξεμβούργο και τι έχουμε πετύχει με την οδηγία του 75. Αρκεί κανείς να έχει μόνο το θάρρος όταν πραγματικά υφίσταται διακρίσεις. Και διάκριση υφίσταται κάποιος μέσα σε μια εταιρεία συγκεκριμένη, όχι σε εθνικό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν και άνδρες στο Λουξεμβούργο. Ας πούμε η κεραμοπία όταν είχαμε τέτοιους κέρδιζαν περισσότερα από εκείνου που ήταν χαλιβουργοί ή ανθρακορίχοι. Αυτό δεν λέει τίποτα λοιπόν σε ό,τι αφορά την οδηγία του 75 πρέπει να πω ότι είναι καλή. Απλώς πρέπει να εφαρμοστεί. Και αν έχετε παραδείγματα όπου δεν εφαρμόζεται η οδηγία, θα πρέπει να προσφεύγετε στα δικαστήρια. Εγώ βοήθησα ε, σε ένα χωριό ε, να γίνουν τέτοιες προσφυγές στη δικαιοσύνη, όπου οι γυναίκες καθαρίστριες πληρωνόντουσαν λιγότερο από καθαριστές και πληρώθηκαν και αναδρομικά γιατί δικαιώθηκαν στο δικαστήριο. 25 εκατομμύρια τότε έπρεπε να τους πληρώσει η κοινότητα, ε, το, το χωριό. Και ήρθαν οι γυναίκες στα γραφεία μου με σαμπάνιες. Και θα ήπιαμε τότε μαζί. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ε, δεν θα τα πω γιατί θα μακρηγορήσω πάρα πολύ και δεν έχουμε χρόνο. Και νομίζω είναι λάθος να λέμε ότι χρειάζεται νέα οδηγία η οδηγία του 1975 που ήμασταν 9 χώρες, αν θυμάμαι καλά, και τώρα είμαστε 27, ε, σε λίγο 28 και δεν πρόκειται να βγει καμία καλύτερη οδηγία. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή που έχουμε. Ε, τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Κοιτάξτε τι κάνει και η Μεγάλη Βρετανία. Αποκλείεται να πετύχετε τίποτα καλύτερο από αυτό που ισχύει τώρα ως κείμενη νομοθεσία από την οδηγία ε, για την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Εάν υφίσταστε ε, διακρίσεις, κινηθείτε, αλλά βασιστείτε σε αυτή την οδηγία. Και ένα τελευταίο για την προστασία των μητέρων. Εγώ δεν υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Γιατί γνώριζα ότι το Συμβούλιο αποκλείεται να τη δεχτεί. Και επίσης, ε, γιατί θεωρούσα ότι την έχουμε παραφορτώσει την οδηγία αυτή. Είναι για τη μητρική προστασία. Αν είχαμε κάνει αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα εδώ και δύο χρόνια θα είχαμε πετύχει μια πρόοδο για τις γυναίκες σε διάφορες χώρες που έχουν μόνο 14 εβδομάδες ε, αδιαμητρότητας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, είναι 16 ε, ε, εβδομάδες, συν τέσσερις όταν θυλάζεις και φυσικά θυλάζουν όλες οι γυναίκες για να πάρουν και ένα μήνα παραπάνω άδεια. Ε, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αλλά την έχουμε παραφορτώ στην οδηγία. Το παρακάναμε. Είπαμε 20 εβδομάδες. Ε, πο πολλές χώρες δεν συμφωνούν γιατί το θεωρούν υπερβολικό. Μετά γιατί το φορτώσαμε, γιατί μιλάμε για γονική άδεια, πατρική άδεια, της Παναγίας στα μάτια. Ταυτόχρονα ήμουν και η συγγήτρια για μια οδηγία για την ίση μεταχείριση των αυτοαπασχολουμένων. Και εκεί πρόκειται για την προστασία των μητέρων και κυρίως για την κοινωνική ασφάλιση. Την έκθεση αυτή την ε, έκανα με τη λογική μου και πάλι δεν επέρασα από το Συμβούλιο, ούτε τους επέβαλα όλα όσα ήθελα, αλλά κατάφερα, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Με τη λογική όταν είμαστε στη συναπόφαση, μπορούμε να κινούμε καταστάσεις. Με τους παραλογισμούς δεν κερδίζουμε τίποτα. Και η έκθεση για την προστασία των μητέρων που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, πραγματικά υπόδειγμα παραφροσύνης και παραλογισμού για το πώς δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη συναπόφαση. Αυτά και σταματώ εδώ. Ε, Σας ευχαριστούμε. Θέλετε... Δεν θέλετε να ακούσουμε και κάποιες άλλες παρεμβάσεις και μετά να απαντήσετε αν δεν σας πειράζει. Η κυρία Εστρέλα παρακαλώ. Ε, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τις ε, συναδέλφους από τη Γερμανική Βουλή και θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση που θέσατε για την επωνομαζόμενη οδηγία για την άδεια μητρότητας. Όντως, ε, πρόκειται για μεγάλη ανησυχία το Κοινοβουλίο μας. Η έκθεση μου εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2010 τον Οκτώβρη και έκτοτε έχει αποτελματωθεί το ζήτημα στο Συμβούλιο. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες που ήδη ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια προφορική ερώτηση παραδείγματος χάρη, προς την Δανική Προεδρία, επιστολές, συσκέψεις με τις διαδοχικές προεδρίες. Α, και θέλω να τονίσω ότι ε, στην Πολωνική Προεδρία καταβάλαμε σημαντικότατη προσπάθεια και συγκεκριμένα έγινε ένα Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων για αυτό το ζήτημα ακριβώς. Και παρόλες αυτές τις προσπάθειες από πλευράς των διαδοχικών προεδριών και του Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ακόμη επίσημα δεν έχει αντιδράσει, δεν έχει τοποθετηθεί το Συμβούλιο. Όσο λοιπόν δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα το Συμβούλιο, είναι αδύνατον να ξεκινήσουμε διαπραγμάτευση. Από πλευράς μας διαθεσιμότητα υπάρχει για έναν άτυπο διάλογο, με τρόπο ώστε να διαπιστώσουμε ποια είναι τα σημεία σύγκλησης και ποια είναι τα σημεία ε, επί των οποίων ε, δεν μπορεί να δώσει σε καμία περίπτωση τη συγκατάθεσή του το Συμβούλιο. Από πλευρά Συμβουλίου δεν υπήρξε καμία εκδήλωση βούλησης ε, διαλόγου επισήμου ή ατύπου. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη που θα ήθελαν να διαπραγματευτούν είναι αντιμέτωπα με άλλα κράτη-μέλη που δεν επιθυμούν την διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη των Εθνικών Κοινοβούλων. Απευθύνω ειδική έκκληση προς τις συναδέλφους ε, ως εκ τούτου σήμερα αν συζητηθεί το θέμα στην Γερμανική Βουλή, να καταλήξετε σε μία θέση και να μας προσφέρετε την υποστήριξή σας. Οποιαδήποτε κίνηση, οποιοδήποτε διάβημο κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτο και κυρίως πολύ χρήσιμο. Το ζήτημα έχει συζητηθεί επανειλημμένο στο Κοινοβούλιο. Ε, οι ψήφισαν με πλήρη επίγνωση των ζητημάτων οι βουλευτέ στην ψηφοφορία και εγκρίθηκε η έκθεσή μου με ευρεία πλειοψηφία. Ξέρουμε πόσο χαλεπή είναι η καιρή που βιώνουμε. Είναι άνευ προηγουμένου η τρέχουσα κρίση. Παρόλα αυτά έχουμε ένα άνοιγμα. Θα μπορούσαμε λόγου χάρη σταδιακά να εφαρμόσουμε τα εν λόγω μέτρα, διότι θεωρούμε πως αυτή η οδηγία 19 ετών είναι παροχημένη ήδη. Δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες των οικογενειών, των παιδιών, των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτό το λόγο θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε, να επιτύχουμε μια βαθμισμένη νομοθεσία. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε να εφαρμοστεί, ξαναλέω, σταδιακά αυτή η νομοθεσία. Ήδη έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση. Λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική Ευρώπη 2020, Παραδεχόμαστε επίσης ότι ο ορίζοντας για την πλήρη υλοποίηση της πρότασης που ενέκρινε το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να τοποθετηθεί το 2020. Για να μην μακρηγορώ, ήθελα μόνο να τονίσω ότι από πλευράς του Κοινοβουλίου Υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα πνεύματος ε, με στόχο να εξευρεθεί μία συνενετική λύση που θα μας οδηγήσει στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Θα θέλαμε επίσης από πλευράς του Συμβουλίου να διαπιστώσουμε το ίδιο άνοιγμα, ούτως ώστε να εκινήσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία ακόμη και άτυπη, εάν αυτό επιθυμεί το Συμβούλιο, ούτως ώστε μεταγενέστερα να καταλήξουμε στην απαιτούμενη για την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας ε, λύση. Ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με την άδεια πατρότητας. Δεν προβλέπεται στην ε, κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία άδεια πατρότητας. Υπάρχει μια οδηγία για την γονική άδεια και υπάρχει και αυτή η οδηγία για την μητρική άδεια. Εμείς ήδη έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εάν αναλάβει μια πρωτοβουλία ή ανακοινώσει την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ε, τρική άδεια. Είμαστε στη διάθεσή της για να αναλύσουμε αυτήν την ε, πρόταση για να καταλήξουμε σε μια νομοθετική ρύθμιση για την άδεια πατρότητας. Πάντως θεωρούμε πώς πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, η άδεια μητρότητας και η άδεια πατρότητας. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπερασπιστούμε την ε, δίκαιη κατανομή των ευθυνών η ευθύνη των παιδιών δεν είναι αποκλειστική για τη γυναίκα. Ο στόχος είναι να προαγάγουμε την ε, συμφιλίωση της ιδιωτικής ε, και της επαγγελματικής ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες του τέστην. Ε, ε, ε υπόψη το ότι ε, η κοινωνία, επιθυμούμε εμείς να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες που αναδύονται από την ίδια την κοινωνία με αυτό τον τρόπο. Καλώς ορίσατε, να πω κλείνοντας το Κοινοβούλιο και να σας συγχαρώ για την εξαιρετική επιτέλεση των καθηκόντων σας στην Επιτροπή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχουμε άλλον, άλλη μια ομιλήτρια και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις απαντήσεις και μετά θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ομιλήτρες. Η κυρία Μπάουερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε. Είναι μεγάλη χαρά που σας βλέπω εδώ. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι στις επισκέπτριές μας. Λοιπόν, πολλά πράγματα υπόθηκαν και δεν συμφωνώ με όλα. Όμως, πρέπει να δούμε ποιες πολιτικές δυνατότητες υπάρχουν. Τι είναι καλό όταν το βλέπει κανείς απόλυτα και θεωρητικά και τι είναι εφικτό μεσοπρόθεσμα. Δεν είναι να δει κανείς μόνο είναι δυνατόν, αλλά και πότε μπορεί να εφαρμοστεί κάτι. Και δεν μπορούμε να τα προβλέπουμε όλα αυτά πάντα επακριβώς. Τι μπορεί να εφαρμοστεί πότε. Λοιπόν, πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την όλη κατάσταση. Όσον αφορά την μητρική άδεια, κάναμε διάφορες ενδιαφέρουσες δοκιμές συλλέξαμε απόψει. Κάθε φορά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ελάχιστε κοινέ προδιαγραφές. Έχουμε τεράστια προβλήματα, διότι ποικίλουν τα συστήματα προνοίας κατά πολύ σε κάθε κράτο μέλο, οπότε είναι δύσκολο να καταρτήσουμε κοινέ προδιαγραφές. Όσον αφορά όμω τη μισθοδολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, μια μικρή διευκρίνηση. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με αυτό που είναι στην ιστοσελίδα του, της Eurostat δείχνει ότι υπάρχει διαφορά της τάξης 16,7% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γενική προσέγγιση είναι αυτή, δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες. Δεν αναφέρονται με μονομένοι τομείς, είναι ένας μέσος όρος μισθών, στον οποίο γίνεται υπολογισμό της διαφοράς. Ε, δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την παιδεία και την κατάρτιση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όσον αφορά τις αμοιβέ υπάρχει αυτή η διαφορά. Πολύ συχνά δεν υπάρχει και διαφορά όσον αφορά την πρακτική εμπειρία ανδρών και γυναικών. Παραμένει όμως η διαφορά στις αμοιβέ. Πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Λούλινγκ. Μπορεί να στραφεί κανείς στη δικαιοσύνη, αλλά υπάρχει διαφορά. στην Ηνωμένο Βασίλειο, Φερρυπίν. δεν υπάρχουν κυρώσεις. Αν απευθυνθεί κανείς στο δικαστήριο, ούτε στη χώρα μας, στη Σλοβακία, για να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να καλύψει τα έξοδα της δίκης. Διερωτηθήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τροποποιήσουμε μια πανάρχια οδηγία του 1975 που αναθεωρήθηκε το 2006. Τι μπορούμε να κάνουμε για να λειτουργεί πραγματικά αυτή η οδηγία. Τι μπορούμε να κάνουμε στις συγκεκριμένε χώρες. Φέτος, εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποσχεθεί να υποβάλει μια πρόταση. Στην πρόταση θα πρόβλεπε τις συλλογικέ δράσεις, class action, προσφυγή συλλογική στα δικαστήρια. Οι συνάδελφοι πρότειναν και σε αυτή την περίπτωση των μισθολογικών διαφορών να υπάρχει δυνατότητα του class action. Είναι αποτελεσματικότατο εργαλείο αυτό. Προσπαθήσαμε να δούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις που τεχνικώς πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν συνολικά για να μειωθεί η μισθολογική διαφορά αλλά για να μην περιμένουμε 100 χρόνια για να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, δεν μπορείτε να απαντήσετε εσεί και μετά θα συνεχίσουμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Λέει ο πρόεδρο, έχετε το λόγο εσεί από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ε, ναι, πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Τώρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε λεπτομερώς σε κάθε μία από τις τοποθετήσεις σας. Κυρία Λούλινγκ, σίγουρα είναι πάντα δύσκολο να βρίσκει κανείς τη σωστή οδό. Και μπορούμε να κάνουμε και ατέρμονες συζητήσεις. Ακριβώς όμως για αυτό το λόγο θεωρώ σωστό να υπάρχουν ποσοστώσεις στα εποπτικά συμβούλια των επιχειρήσεων. που δεν είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της καθημερινής διοίκησης των επιχειρήσεων, <laughs> αλλά είναι ένα άλλο όργανο εποπτείας της επιχείρησης. Και θα πρέπει να δείξουμε ε, ότι ανεξάρτητα από τη μορφή που έχουν σε κάθε κράτος μέλος, αυτά τα όργανα, τα εποπτικά των επιχειρήσεων και όχι το Διοικητικό Συμβούλιο, ε, είναι κάτι ξεχωριστό μέχρι τώρα κυριαρχούνται, από ανδροκρατούνται. Και έχουμε ευθύνη και ε, πανευρωπαϊκά αλλά και στη χώρα μου την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι κατοχυρωμένο στο θεμελιώδη νόμο, στο σύνταγμά μας ότι προάγουμε την ισότητα των φίλων. Έχουμε καθήκον να το πράξουμε. Και αν σε αυτά τα επίπεδα άσκησης, επιρροής αλλά και εξουσίας παραμένει μηδενική ή σχεδόν μηδενική παρουσία των γυναικών και η εικόνα τους, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι οι γυναίκες δεν έχουν την ε, που τους αναλογεί λόγω της μόρφωσης ή των δυνατοτήτων τους. Γι' αυτό υποστηρίζω και το θέμα των ποσοστώσεων, παρόλο που έχω ε, συνηθίσει από μακρά πολιτική εμπειρία να ε, ενεργώ με σύνεση, σίγουρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και μια κίνηση. Και ελπίζω να γίνει αυτό και από τη Γερμανική Βουλή και υπάρχουν και συντηρητικές γυναίκες που έχουν αρκετή ε, τόλμη για να μπουν σε αυτή την ατραπό. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουν και το θάρρος και το στένος να το επιβάλλουν αυτό θα πρέπει να είμαστε ενωμένε όλες οι γυναίκες, να έχουμε ε, υποστήριξη των αδρών και να καταλάβουμε την αξία αυτών των θεμάτων. Τώρα, για το θέμα ε, των μισθολογικών διαφορών, θα πρέπει να ε, συγκρίνουμε συγκρίσιμα μεγέθη μεταξύ τους. Δεν έχει λυθεί το θέμα, παραμένει ζήτημα και ακούω και από νέε γυναίκες τι λέγουν για τον πρώτο μισθό που είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο καν τον διαπραγματεύονται από ό,τι συνηθίζουν οι άντρες. Ιδιαίτερα όταν έχουν και οικογένεια και δεν κάνουν αποκλειστικά καριέρα ή επαγγελματική ε, δραστηριότητα. Και οι γυναίκες χρειάζεται να απολογούνται κιόλας που έχουν οικογένεια. γιατί αυτό δεν θεωρείται εργασία και ε, τελικά τις ξεγελάνε, τις ε, ε, ε μειώνουν, τις υπονομεύουν και δεν τις πληρώνουν ως θα όφυλαν. Παρόλο που οι γυναίκες εργάζονται στην οικογένεια και ουσιαστικά έχουν διπλή επιβάρηση και δεν θα πρέπει, όχι, μόνο θα πρέπει να πληρώνονται λιγότερο, αλλά πληρώνονται περισσότερο από τους άνδρες που είναι σε ανταγωνισμό μαζί τους για την οδηγία για την προστασία των μητέρων. Και εγώ θεωρώ ότι είναι υπερφωτωμένη και είμαι φιλελεύθερη, έχουμε την ίδια αντίληψη σε αυτό. Και θα πρέπει να την ξανασκεφτούμε οπωσδήποτε επί της αρχής ξανά. Α, απευθύνομαι με αυτά και στις άλλες συναδέλφους, όχι μόνο στην κυρία Λούλινγκ. Νομίζω άρχισα να απαντώ στην κυρία Λούλινγκ, αλλά αφορά όλες τις υπόλοιπε τοποθετήσεις, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την ευκαιρία που μας δίνετε και πάλι να συμμετάσχουμε σήμερα εδώ. Και εγώ έχω την ίδια εμπειρία με τη συνάδελφο από το Λουξεμβούργο. 40 χρόνια πολιτική ισότητας κάνω κι εγώ, αλλά 40 χρόνια ε, πολιτική ισότητας ε, έχει κάνει προόδους σε ρυθμούς σαλιγκαριού και το θέμα της ίσης αμοιβή ανδρών και γυναικών θα πρέπει να είναι κάτι το προφανές και αυτονόητο. Γι' αυτό έτσι χάνω λίγο την υπομονή μου σε αντίθεση με εσά ίσως, γιατί μετά από 40 χρόνια χωρίς συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα δεν έχουμε προχωρήσει ούτε βήμα. Τις εθελούσιες ρυθμίσεις τις έχουμε ζήσει δυστυχώς στη Γερμανία. Το κάναμε αυτό, κάναμε και συμφωνία στη Γερμανία, οι επιχειρήσεις και η πολιτική ε, ότι θα αλλάξει λέει κάτι στην πολιτική ισότητας και μετά από 11 έτη η συμφωνία αυτή δεν οδήγησε πουθενά. Ε, όχι μόνο δεν ε, έγιναν βήματα προς τα εμπρός, αλλά και οπισθοδρομήσεις έγιναν. Η οδηγία είναι το σωστό μέτρο και για την ίση αμοιβή και για τις ποσοστώσεις. Μόνο με νομοθετικό μέτρο γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε πια να ε, ανεχόμαστε να διαδηλώνουμε κάθε χρόνο και να απαιτούμε ίση αμοιφή. E το ξέρω ότι είναι μεσιόρι. Ε, ε, αυτό είναι το σκάνδαλο όμως, ότι ο μέσος όρος δείχνει ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ακόμα η διαφορά. δηλαδή, σε θέσεις διευθυντικές, αυτό το 16-17% μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Στη Γερμανία δεν μέχρι το 35%. Εμείς ως γυναίκες δεν μπορούμε να τα ανεχόμαστε πλέον αυτά, ότι να αξιολογείται η δική μας εργασία χειρότερα από εκείνη των ανδρών. Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την αξίωση, χρειαζόμαστε και ένα δρόμο προς μια οδηγία που να είναι πιο δεσμευτική στην Ευρώπη. Η δική σας πρόταση μου άρεσε πολύ, κυρία Μπάουερ, για τις ε, ε, συλλογικές αγωγές. Δηλαδή, να μην πηγαίνει ο καθένας στο δικαστήριο ατομικά, γιατί δεν το κάνει. Γιατί φοβάται κιόλας μην τον απολύσουν, μην την απολύσουν. Αλλά να έχουμε μια συλλογική δράση έτσι με συλλογικές αγωγές ή κάτι τέτοιο έτσι ώστε να μην απολύονται οι εργαζόμενες αν προσφεύγουν στα δικαστήρια μεμονωμένα. Καλή ιδέα, αλλά θα πρέπει να είναι πιο δεσμευτικά όλα αυτά για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Άλλες τρεις ομιλήτρες έχουμε. Σένισιν, Κιβίτ και Μουρβάη και στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να παρεμβετε εκ νέου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, θέλω να πω κάποια πράγματα που καμιά φορά τα ξεχνάμε. Οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες δεν αντιβαίνουν πουδενή τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Αντιθέτως, χρειάζονται για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία της αγοράς. Σήμερα υπάρχει σημαντική αντίσταση όσον αφορά το διορισμό γυναικών σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Διότι έτσι ήταν πάντα η αγορά. Ταυτόχρονα έχουμε ποσοστώσεις, ειδικέ ποσοστώσεις για τους άνδρες. Στην Πολωνία αυτές οι ποσοστώσεις φτάνουν το 90% όσον αφορά τα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και για, σε κάποιες περιπτώσεις πάει και 98% και δεν είναι κάτι που αντιβαίνει ε, το σεβασμό των ανδρών, την ευφυΐα των ανδρών και δεν ενοχλούνται οι άντρες καθόλου. Ενώ οι γυναίκες ε, υποτίθεται πρέπει να αισθάνονται άσχημα αν η ποσόστοση φτάνει 40-50%. Σύμφωνα μια έρευνα, αν υπήρχε ποσόστοση για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 5 με 7%. Διότι οι γυναίκες διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο τις επιχειρήσεις από ότι οι άντρες. Αναλαμβάνουν λιγότερους κινδύνους οι γυναίκες. Οπότε, αν ειχαμε μισό 50-50 γυναίκες και άντρες ε, στα διοικητικά συμβούλια, θα λειτουργούσαν πιο ορθολογικά οι εταιρείε από ότι όταν υπάρχουν περισσότεροι άντρες στα διοικητικά συμβούλια. Αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες, βέβαια, ούτε αυτό θα ήταν καλό. Ταυτόχρονα, όταν οι πρόεδροι εταιριών είναι, διορίζονται μάλλον πρόεδροι εταιριών, ακόμα και αν οι γυναίκες έχουν καλύτερη παιδεία και ικανότητες, διορίζονται οι άντρες παρόλα αυτά. Διότι η αλλαγή του Προέδρου επηρεάζει τις μετοχές της επιχείρησης. Μπορεί, όταν γίνεται η αλλαγή πέφτουν κατά 2% οι μετοχές. Αν διοριστεί γυναίκα, οι μετοχές πέφτουν κατά 4 με 5%. Οπότε και αυτό είναι άλλη μια ένδειξη να λάβετε υπόψη ότι είναι καλύτερο να αγοράζει κανείς μετοχές εταιριών που έχουν γυναίκα, νέα γυναίκα πρόεδρο, διότι μετά από μια περίοδο οι μετοχές θα ανέβουν και πάλι. Και δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών που χειρίζονται οι άντρες και οι γυναίκες. Αυτά θα πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε συνεχώς, διότι αυτή η έρευνα, αυτά που σας είπα, το λησμονείται συχνά. Ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα την κυρία Κλειβέτη. Σύντομα. Α, συγγνώμη. Θα ήθελα να πω μόνο σύντομα ότι στις 11 παρα 10 πρέπει να φύγουμε διότι έχουμε ραντεβού επόμενο στη συνέχεια. Okay. Okay, I didn't know that. I thought we had the time to 11, so. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε μέχρι τις 11, είχα καταλάβει. Καλά, ας ακούσουμε την κυρία Κλειβέτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω τις συναδέλφους από την Bundestag. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο θέματα σημαντικότατα για μένα. Να σας πω τι διάβασα κάπου. Λοιπόν, αν το όνομα μιας τράπεζας που δημιούργησε την κρίση ήταν Lehman Sisters και όχι Lehman Brothers, τότε δεν θα υπήρχε κρίση. αναφέρθηκε. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά Υπάρχουν τέτοιες απόψεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άντρες αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους από τις γυναίκες. Ε, όσον αφορά τις ποσοστώσεις και τη μέρημνα της Επιτρόπου Ρέντινγκ να εισαγάγει ποσοστώσεις για διοικητικά συμβούλια τραπεζών και επιχειρήσεων, αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τις γυναίκες. Προσωπικά, θα ήθελα να δω γυναίκες σε όλους τους φορείς λήψεως αποφάσεων σε θέσεις υπεύθυνε. διότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία όσον αφορά τις εργασίες που κάνουν άντρες και γυναίκες. Σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Μπάουερ, οι εθνικές πρακτικές και διάφορα μεμονωμένα παραδείγματα εθίγησαν Οπότε θα αναφέρω και εγώ κάτι. Στη Ρουμανία, στην πατρίδα μου, ε, έχουμε γονική άδεια για δύο χρόνια που δίνεται για τα παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Δεν υπάρχει αναλλακτική για τις Ρουμάνες γυναίκες. Νωρίς στην καριέρα τους οι γυναίκες μπορούν να αποφασίσουν να πάρουν άδεια διετή. Υπάρχουν διχασμένες απόψεις από αυτού. Αλλά κατά την άποψή μου το κράτος πρέπει να επενδύει περισσότερα για τις οικογένειες, να βοηθά τις οικογένειες, να ενθαρρύνει τη μητρότητα, ε, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας τα παιδιά να πηγαίνουν σε ε, βρεφικούς σταθμούς, νηπιακούς σταθμούς. Όσον αφορά τη διάρκεια της άδειας νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια ομοιόμορφη λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ σύντομα, ε, έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ, έχουμε ελάχιστο χρόνο, οπότε έχω ένα ερώτημα που έχω, θέλω να θέσω στις επισκέπτριές μας από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε λοιπόν ότι μιλάμε για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την αλληλεγγύη μεταξύ γυναικών. Όταν μιλάμε για τις ε, γερμανικές τοποθετήσεις, τη γερμανική κατάσταση, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι συνθήκες που επικρατούν εκεί είναι διαφορετικές. Η Γερμανία στην πράξη ε, κάνει απικίες, οικονομική απικία την Ουγγαρία και είναι θλιβερές συνθήκες που επικρατούν στην Ουγγαρία. Μόνο 300 ευρώ ε, καταβάλλονται ω αμοιβέ των γυναικών στην Ουγγαρία σε επιχειρήσεις γερμανικές. Αυτό σημαίνει πλήρη στέρηση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αν παράδειγμα χάρη η γυναίκα, μια γυναίκα πρέπει να πάει στο γιατρό, έχει πρόβλημα διότι πολύ συχνά χάνει τη θέση εργασίας της. Το σκεφτήκατε αυτό. Μήπως θα ήταν καλό από πλευράς δικής σας να στείλετε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας της Bundestag στην Ουγγαρία να δείτε τι γίνεται. Σας κάνω επίσημη πρόσκληση και ρωτώ, ξέρετε ότι η Ουγγαρία που είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πάρα πολλές γυναίκες που μεταναστεύουν προς τη Γερμανία και εργάζονται σε πολύ κακές συνθήκες, είναι πολύ συχνά πτυχιούχες που πηγαίνουν να εργαστούν σαν καθαρίστριες ή καμιά φορά καταλήγουν και στην πορνεία. Είναι θύματα του εμπορίου λευκής αρκός. Ε, αυτό αντιβαίνει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις πολύ συχνά μετεγκαθίστανται στην Ουγγαρία και μεταχειρίζονται ουσιαστικά σαν σκλάβους τους Ούγγρους, δίνοντάς τους γελίες αμοιβέ ε, με πολλές στερήσεις. Αντίθετα, αυτό για μας σημαίνει ότι οι πολίτες μας πρέπει να πάνε στη Γερμανία και πάνε με πολύ καλά προσόντα και εργάζονται σε θέσεις που δεν ταιριάζουν καθόλου στην παιδεία τους. Τι σκέφτεστε εσείς γι' αυτά. θα πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις της ε, κρίσης ε, για τις γυναίκες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ή ίσως όχι τόσο στη Γερμανία, αλλά σε άλλες χώρες σίγουρα είναι τεράστιο αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω αν έχετε όμως κάποια σύντομα σχόλια. Το ξέρω ότι υπερβήκαμε αυτό το 11 παρα 10 που μας είπατε, αλλά μπορεί παρόλα αυτά να θέλετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις προστασία των μητέρων και τέτοια ζητήματα, η γονική ε, άδεια ή ο χρόνος ε, των γονέων, όπως είπε η συνάδελφος από τη Ρουμανία, είναι κάτι που ελέγχουμε συχνά ε, στη Γερμανική Βουλή, εάν ανταποκρίνονται και ακολουθούν τις εξελίξεις της κοινωνίας. Στο μεταξύ, εργάζονται πολλές μητέρε. Στη Γερμανία αυτό στο παρελθόν δεν ήταν τόσο συνηθισμένο, γιατί όταν είχαν παιδιά σε προσχολική ηλικία δεν εργάζονταν οι γυναίκες και, έχουμε πρόβλημα στη φύλαξη των παιδιών και σε βρεφονιπιακούς σταθμού. Τώρα, αυτό που ρώτησε η συνάδελφος από την Ουγγαρία δείχνει ότι οι συνθήκε διαβίωση όσο και εργασία των γυναικών στην Ευρώπη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εγώ είμαι δικηγόρος και ακούω τα σχόλια ε, για την κατάσταση των ε, ε, γυναικών της Ουγγαρίας και υπό το πρίσμα της προστασίας της εργασίας των γυναικών στην Ουγγαρία. Δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα, τα νομικά, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ανταλλαγή απόψε και Τώρα είμαστε, είμαστε καθόμαστε σαν αμένα κάρβουνα. Αλλά πρέπει να φύγω και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δεν ανήκω σε εκείνους τους βουλευτές που ε, υπεκφεύγουν και με ασαφείς ε, απαντήσεις θέλουν να αποφύγουν να, να απαντήσουν. Ε, τώρα, σε δύο εβδομάδες, είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στις Βρυξέλλες, ξέρουμε ότι δεν έχουμε χρόνο όλοι, ε, πολύ θα ήθελα να επαναλάβω την πρόσκλησή μου ρητά. Όποιος συνάδελφος ε, θέλει να έρθει ε, είναι ε, ευπρόσδεκτος, προσκεκλημένος. Πραγματικά με εξέπληξε το κλίμα της συζήτησης. Ήταν πάρα πολύ ειλικρινές και πάρα πολύ ανοιχτό και χρειαζόμαστε σίγουρα και άλλες ανταλλαγές τέτοιες απόψεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση χαρήκαμε ιδιαίτερα που σας είχαμε εδώ. ε, ίσως θα υπήρχε δυνατότητα να σε επισκεφτούμε ολόκληρη η Επιτροπή, με κάποια μέλη της Επιτροπής. Ε, όπως είπα και στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια τακτική επαφή, να έχουμε επισκέψεις. Ε, βεβαίως, πάντοτε υπάρχουν περιορισμοί στο χρόνο και θέλουμε όλοι να πούμε τόσα πολλά και δεν προλαβαίνουμε. Πάντως, ε, μεταφέροντας τις σκέψεις μας, δημιουργούνται και διαμορφώνονται οι απόψεις. Αυτή είναι μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Πάντως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Eh, eh, Ωραία, ας περάσουμε τώρα στο σημείο 11. Εξάλληψη των ε, συνδεωμένων με το φύλλο στερεοτύπων στην Ένωση. Δυστυχώς ε, η συγγήτρια, η κυρία Λιωτάρ, ε, ασθενεί σήμερα και δεν μπορεί να έρθει για τη συζήτηση. Υποσχέθηκα να διαβάσω εγώ ένα μήνυμα από πλευρά τη και αν υπάρχουν σχόλια θα τα σημειώσουμε, σίγουρα θα υπάρχουν δηλαδή, θα τα σημειώσουμε ούτω ώστε να ε, περάσουμε προς την κυρία Λιωτάρ το μήνυμά μας ε, για να συνεχίσει εκείνη τις εργασίες της. Ε, θα σας διαβάσω αυτά που μου έδωσε η Κατίκα. Στα αγγλικά μου έδωσε το κείμενο. Θα το διαβάσω στα αγγλικά γιατί είναι δύσκολο να διαβάζω αγγλικά και να μιλάω σου ειδικά. Οπότε θα το διαβάσω στα αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω Όλου του συναδέλφου που υπέβαλαν τόσες πολλές τροπολογίες ως επιτοπλίστων ακολουθούν την, τον ίδιο προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτή μια ευρεία συνένεση στην Επιτροπή των Γυναικών για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά θα προτείνω συμβαστικέ ε, λύσει για να είναι και πιο ευανάγνωστο το κείμενο. Πολλέ ε, τροπολογίε, ε, όπω είπα ακολουθούν τον ίδιο προσανατολισμό και θέλω να αποφύγω τις επικαλύψεις και τι επαναλήψει. Θα υποβάλω κάποιες συμβαστικέ προτάσεις για να συμπεριλάβω και τις ε, ιδέες σας, ε, όχι αποτυπώνοντα βεβαίω την ακριβή διατύπωση που θα εισηγηθείτε εσείς, ελπίζω να το δεχτείτε. Την επόμενη Δευτέρα έχουμε προγραμματίσει συνεδρίαση των συντονιστών από τις 4 μέχρι τις 5 στο 1G1. θα έχουν κυκλοφορήσει τα σχέδια των συμβαστικών τροπολογιών και θα τις συζητήσουμε στην ε, συνεδρίαση αυτή. Στη συνέχεια θα έχουμε στη διάθεσή μας δύο εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε. Ελπίζω να ε, καταλήξουμε σε μια ευρέως αποδεκτή και πλήρη έκθεση. Η δούλη, ο Πρόεδρος, ε, λίγη τώρα το μήνυμα που ήθελε να μας διαβιβάσει η κατοίκα. Θα ήθελα τώρα να αρχίσει η συζήτηση. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν παρατηρήσεις ε, θα, τα, ε, τις ε, σημειώσουμε και θα τις διαβιβάσουμε στην κατοίκα. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε τον λόγο. Η κυρία Τσέσκοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι πάρα πολύ που η κυρία εισηγήτρια απουσιάζει. Αλλά τι να κάνουμε, είναι μες στη ζωή και αυτά. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την έκθεσή της. Έχω κάνει και εγώ μερικές τροπολογίες. Και τώρα και με το μήνυμα που μας έστειλε είπε και η ίδια ότι θα κάνει συμβιβαστικές προτάσεις. Γενικά συμφωνούμε για αυτά τα στερεότυπα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το φύλλο. Και συμφωνώ όλες τις πολιτικές ομάδες. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα μου και πρέπει να πω ότι υποστηρίζω τις περισσότερες τροπολογίες. Ορισμένες από τις τροπολογίες αυτές θα τις στηρίξω όλους ιδιαίτερως Ας πούμε, ένα από τα θέματα που με ενδιαφέρουν είναι η βία με βάση το φύλλο. Και πιστεύω ότι αυτά τα στερεότυπα ε, ε περί το φύλλο οδηγούν σε ανισότητες ε, και στη μεταχείριση. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που θεωρεί ότι έχει περισσότερα δικαιώματα. Οπότε υποστηρίζω αυτές τις τροπολογίες. Ε, ε, στη συνέχεια, πρέπει να σας πω ότι υποστηρίζω και τις τροπολογίες ε, κατά των διακρίσεων και του διαχωρισμού στους χώρους εργασίας. Εδώ τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν και τέτοια μέτρα στη στρατηγική τους και στην νομοθεσία τους και εμείς να έχουμε μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τα επαγγέλματα που εργάζονται, όπου μάλλον εργάζονται σήμερα λιγότερες γυναίκες. Θα πρέπει οι γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο και στο πολιτικό γίγνεσθε και ε, κυρίως τα κράτη-μέλη να υποστηρίζουν τις γυναίκες για να μπορούν να φτάνουν μέχρι τις διευθυντικές σχέσεις, θέσεις συγγνώμη, ή και ηγετικά πόστα στην πολιτική. Επίσης λυπάμαι που δεν είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην προηγούμενη συζήτηση. Άκουσα μερικές ε, τοποθετήσεις και απαντήσεις. Παρακολουθούσα στο διαδίκτυο τη ε, συζήτηση ωστόσο. Και πρέπει να σας πω το εξής. Πριν από 10 χρόνια θα είχα προσυπογράψει λέξη προς λέξη αυτά που είπε η κυρία Λούλινγκ, που μίλησε για λογική προσέγγιση. Αλλά μετά από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί είμαι μητέρα δύο παιδιών, Έχω ζήσει στο πετσί μου αυτέ τι διακρίσεις. Και ο πατέρας των παιδιών μου βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης και με κατηγορεί και κάνει ολόκληρη εκστρατεία γιατί ε, συνέχισα να ε, δραστηριοποιούμε στην πολιτική ε, αφού το απέκτησα τα παιδιά μου. Λοιπόν, υπάρχουν στερεότυπα, τα έχω ζήσει εγώ στο πετσί μου και πρέπει να τα, τα πολεμήσουμε. Αυτό αφορά και την προβληματική των ποσοστώσεων που επίκειται τώρα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να το συζητούμε καν αυτό το θέμα. Η κοινωνία ολόκληρη, συμπεριλαμβανομένων και των ανδρών, πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αυτό είναι ο στόχος το κάτω-κάτω. Ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να επιβάλλουμε νομοθετική ρύθμιση, την οποία πρέπει να σας πω δεν ε, πρεσβεύω 100%. Αλλά η κυρία Ρέντινγκ, η Επίτροπος, είναι πάρα πολύ θαραλέα και έχει βάλει τόσο υψηλού στόχους ε, που αξίζει να υποστηριχθεί. Και είναι καλό και μόνο το γεγονός ότι θα συζητούμε πια αυτά τα θέματα. Διότι κάθε φορά που υποχρεώνεται μια γυναίκα να επιλέξει ε, εργασία ή οικογένεια, ε, βρίσκεται σε μια σύγκρουση. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία οι κοινωνίες. Τα είπαν οι συνάδελφοι από τη Γερμανική Βουλή αυτά. Να μην έχει την αίσθηση η γυναίκα ότι θα πρέπει να απολογείται και όλες να ζητάει συγγνώμη από την κοινωνία ότι ε, εργάζεται και έχει και οικογένεια. Πολύ ωραία τα είπανε οι Γερμανίδες ε, βουλευτές. Και εγώ τα, αυτά τα προσυπογράφω τώρα μετά από τη δεκαετή μου εμπειρία. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση που συζητούμε τώρα. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λιωτά. Υπάρχει πραγματικά έδαφος ε, για να προχωρήσουμε γιατί συμφωνούμε όλες οι ομάδες. Κυρία Νικολάη, τώρα ε, θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Λεωτάρ για αυτή την έκθεση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δυστυχώς όμως είμαστε υποχρεωμένες να ξανασυζητήσουμε τα στερεότυπα αυτού τον αιώνα. Είναι δύσκολο αυτό για μας, διότι είναι σημαντικό το εξής ερώτημα. Πώς μπορούμε να διδάξουμε στους άλλους τις βέλτιστες πρακτικές στις γυναίκες παραδείγματος χάρη που έχουν ανεμιχθεί στην Αραβική Άνοιξη πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό δεν εφαρμόζουμε σωστά στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα των φύλων αυτή η αιμονή των στερεοτύπων με βάση το φύλλο είναι μεγάλο πρόβλημα οι διαφορές των αμοιβών, η συζήτηση για τις ποσοστώσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι ε, αποτελέσματα αρνητικών στερεοτύπων που δημιουργούνται όσον αφορά τις γυναίκες. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα ακούμε ότι δεν υπάρχουν, ε, αυτή δεν είναι δουλειά για τη γυναίκα, αυτό δεν είναι ζήτημα για τη γυναίκα, δεν είναι θέση της γυναίκας αυτή. Και ακούμε και άλλες αποθαρρυντικές φράσεις που αποθαρρύνουν τις νέες γυναίκες να ζητήσουν να καλύψουν Κάποιε θέσει σαν μηχανική, σαν ειδικέ για την πληροφορική κλπ. Ένα σημαντικό θέμα που αναφέρεται στην έκθεση είναι τα σχολικά προγράμματα, το πρόγραμμα των μαθημάτων. Και εκεί έχουν εισβάλει τα στερεότυπα με βάση το φύλλο. Διαμορφώνεται το σχολικό πρόγραμμα και διαμορφώνεται ο τρόπος με τον οποίο το αγόρι το κορίτσι βλέπει τον εαυτό του. Και αυτό διονύζει την ανισότητα στις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Ε, μπορώ να αναφέρω μία βέλτιστη πρακτική που θεωρώ που έχει σαχθεί όταν ήμουν υπουργό ε, για ισότητα των φίλων στη χώρα μου. Υποχρεωτική συμπερίληψη του θέματος των φίλων για τους δασκάλους. Να διδάσκεται πρώτα ο δάσκαλος για την ισότητα των φίλων για να αποφεύγεται η δημιουργία στερεότυπων και μετά ο δάσκαλος ή η δασκάλα να διδάσκει σωστά τα παιδιά. Το τελευταίο που θεωρώ σημαντικό είναι τα ΜΜΕ ε, που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Είναι πολύ ισχυρό μέσο και εδώ επικρατούν πολλά στερεότυπα. Η τροπολογία μου υπογραμμίζει τη σημασία συμπερίληψης αγοριών και ανδρών στην διαδικασία λήψης υπόψη της διάστασης ισότητα των φύλων σε όλου του τομεί. είναι σημαντικό βήμα αυτό. Δεν αρκεί, αλλά σημαντικό βήμα. Ε, αν μπορούμε να το πούμε ότι η έκθεση είναι μία έγκαιρη προειδοποίηση για αυτό το πρόβλημα. Πολύ καλή ιδέα να επιλεχθεί μια τέτοια έκθεση για να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για το θέμα αυτό. Ότι παραμένουν αυτές οι νοτροπίες, αυτά τα στερεότυπα στην κοινωνία. Ε, υποστηρίζουμε πλήρως την έκθεση από πλευράς της ομάδας της Άλντε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Ε, Υπάρχει κάποιο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι. Καλά, άμα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω μόνο ότι στις 6 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή και κατά πάσα πιθανότητα το Μάρτιο του 2013 θα περάσει το θέμα από την Ολομέλεια. Ολοκληρώνεται το σημείο και παίρνουμε τώρα στο 12. Η ένταξη των μεταναστών, οι συνέπειε στην αγορά εργασία, καθώ και η εξωτερική διάσταση του συντονισμού τη κοινωνική ε, ασφάλιση, ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ακούσουμε την κυρία Σένιτσιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, έχετε ένα σχέδιο γνωμοδότησης μπροστά σας, όπου εκεί συμπεριλαμβάνω τις σημαντικότερες πτυχές όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Όμως, περιορίστηκα πολύ από τον αριθμό των ε, λέξεων που μπορούσα να χρησιμοποιήσω στο έγγραφο δεν μπορούσα να συμπεριλάβω όλα όσα ήθελα και γι' αυτό ήδη ετοίμασα κάποιες τροπολογίες που θα υποβάλω για την γνωμοδότησή μου. Εγώ είμαι ανοιχτή σε προτάσεις σας και είμαι ευγνώμων που μπορώ να ασχοληθώ με το θέμα. Η μετανάστευση των γυναικών ήταν πάντα σημαντικό τμήμα της μετανάστευσης εν γέννη. Είναι πάνω από 50% των μεταναστών στην Ευρώπη οι γυναίκες είναι πολύ σημαντικές οι γυναίκες σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα είδη των, της μετανάστευσης. Ε, κατά το παρελθόν, κυρίως οι άντρες έψαχναν μια καλύτερη ζωή και οι γυναίκες ερχόταν μόνο σαν σύζυγοι, σαν σύντροφοι. Ε, γι' αυτό πολύ συχνά ε, έμεναν στο περιθώριο γυναίκες όσον αφορά την νομοθεσία. Δεν ήταν στο επίκεντρο της νομοθεσίας ε, τώρα οι περισσότερες γυναίκες που έρχονται στην Ευρώπη ε, θέλουν να έρθουν εδώ για λόγους οικονομικούς, θέλουν να εργαστούν σε πολλά επαγγέλματα που κυριαρχούνται από τις γυναίκες και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα στερεότυπα που υπάρχουν σαν αυτά τα Έρχονται να εργαστούν οι γυναίκες στον τομέα του καθαρισμού, καθαρισμού συγγνώμη, ε, διασκέδασης, γαστρονομίας ε, όμως θα έλεγα ότι όσο αφορά τη διασκέδαση περισσότερα αυτά ταιριάζουν, ε, εντάσσονται κοντά στην πορνεία. Πολύ συχνά είναι παράνομε οι θέσεις ε, εργασία αυτές που καλύπτουν και ακόμα και αν είναι νόμιμα, εργάζονται νόμιμα, παρόλα αυτά έχουν, δίνουν πολύ, τους δίνουν πολύ άσχημα συμβόλαια, πολύ κακές συνθήκες εργασίας, ασφάλιση κλπ. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα όσον αφορά τη σωστή εφαρμογή των πολιτικών είναι ότι βλέπουμε τους ε, μετανάστες από τη σκοπιά των ανδρών. Οι μετανάστες θεωρούμε ότι αν υπάρχει μια οικογένεια εξαρτώνται πολύ από τον άνδρα. Οπότε υπάρχει διάκριση κατά των γυναικών μεταναστριών. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε κάποιες, ε, να ενισχύσουμε τις γυναίκες, τις μετανάστριες, να μάθουν ότι έχουν δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα οι μετανάστριες και θα πρέπει να τις προστατεύουμε κατά ιασδήποτε παρενόχλησης, κατάχρησης, διακριτικής μεταχείρισης. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι μετανάστρες ε, είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα. Είναι διαφορετική κατηγορία και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουν στρατηγικές των χωρών υποδοχής κάτι που λειτουργεί για μια ομάδα γυναικών δεν λειτουργεί απαραίτητα για μια άλλη ομάδα γυναικών. Το σημαντικότερο για μια επιτυχή ένταξη των μεταναστριών είναι το εξή κατά την άποψή μου. Ανεξάρτητο νομικό καθεστώς. Πολλές μετανάστριες δεν μπορούν να εργαστούν διότι δεν υπάρχουν νομικές δυνατότητες για να εργαστούν. Αυτές που ζητούν άσυλο δεν μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε δουλειά. Οι περισσότερες μένουν ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας και μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν μια θέση εργασίας. Πολλές παράνομες μετανάστριες εργάζονται σαν babysitter ή σαν ε, καθαρίστριες και δεν έχουν δικαιώματα. Ε, πρέπει επιπλέον να αναγνωρίσουμε και την παιδεία τους, τα προσόντα τους παρά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν πολιτικές υποστήριξης των μεταναστριών και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μετανάστριες να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους στην αγορά εργασίας. Δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αφορά τις διαδικασίες για την αναγνώριση πτυχίων Φερρυπίν. Και ακόμα και αν λάβουν τις πληροφορίες, αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες ε, και υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Πολλές γυναίκες παρετούνται ευθύ εξ αρχής από την όλη προσπάθεια και δέχονται απλώς θέσεις με χαμηλή αμοιβή, θέσεις που απαιτούν ελάχιστα, ε, ελάχιστα προσόντα στη μαύρη αγορά εργασίας. Πολύ συχνά υποτιμώνται, υποτιμώνται τα προσόντα τους και πέφτουν θύμα ε, της πατάλης εγκεφάλων όπως αποκαλείται. Πολλές μετανάστριες εργάζονται σε θέσεις που υπολείπονται κατά πολύ των προσόντων τους θα πρέπει να εστιαστούμε επί του συστήματος αναγνώρισης των, των προσόντων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες και αν κάποιος έρθει ανειδίκευτος θα πρέπει να τύχει υποστήριξης για παιδεία, για κατάρτιση, για να βρει μια δουλειά στη χώρα υποδοχής. Παροχή υπηρεσιών λοιπόν για την αγορά εργασίας. Πρέπει να προσφέρουμε σε αυτές τις γυναίκες πληροφορίες όχι μόνο για τις προσφορές θέσεων απασχόλησης αλλά για το εργατικό δίκαιο, για τις διαδικασίες, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με διάφορους οργανισμούς και θεσμούς που ίσως να, θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, να τις βοηθήσουν. Χρειάζονται επίσης συμβουλές όσον αφορά ε, την αντιμετώπιση κακών συμπεριφερών κατά ε, παρενόχληση, κατάχρηση ε, και η γλώσσα είναι πρόβλημα. Αν ε, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα τη χώρα υποδοχή, μπαίνουν πολύ συχνά στο περιθώριο, βγαίνουν εκτό τη αγορά εργασία και δεν έχουν πολλέ κοινωνικέ επαφέ. Πολύ συχνά οι άντρε και όχι οι γυναίκε μαθαίνουν γλώσσε. Και έτσι δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο. Επειδή οι γυναίκε δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, δεν αισθάνονται ότι έχουν ένα κίνητρο να ψάξουν να βρουν δουλειά και δεν ψάχνουν να βρουν δουλειά διότι δεν ξέρουν τη γλώσσα και επιπλέον πολύ συχνά θα πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους και ίσως κάποιες από αυτές δεν έχουν οικονομικούς πόρους που τους απομένουν για να προσπαθήσουν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα για να μάθουν μια γλώσσα. Άλλο πρόβλημα είναι η ένταξή τους σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Θα έπρεπε να συντονιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση τέσσερους πυλώνες. Ίση αντιμετώπιση, να μην υπάρχει διάκριση, ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας, Τα κεκτημένα δικαιώματα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης και η ασφάλιση, ο χρόνος ασφάλισης και οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να αναγνωρίζονται στη χώρα υποδοχής. Βέβαια γνωρίζω ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών η νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές διαφορές. Και είναι δύσκολο επίσης να αναλυθούν τα διάφορα συστήματα και τα 27 συστήματα, διότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των γυναικών που εμπλέκονται σε αυτά τα κοινωνικά συστήματα, πόσε από αυτές είναι μέσα στα κοινωνικά συστήματα. Οι περισσότερες μετανάστριες δεν γνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να δικαιούνται ε, να λάβουν κάποια επιδόματα και πολύ συχνά δεν έχουμε διμερεί συμφωνίες με τις τρίτες χώρες, οπότε δεν μπορούν να μεταφέρουν τα δικαιώματά τους, τα συνταξιωτικά δικαιώματά τους ή άλλα κοινωνικά δικαιώματα στη χώρα υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτονται καθόλου αν του συμβεί κάτι. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι με πολλή γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία είναι τεράστιο εμπόδιο για τις επαφές με τη δίκηση κυρίως όταν μιλάμε για τα συστήματα κοινωνικής ε, ασφάλισης. Αυτά λοιπόν είναι μόνο κάποιες πρώτες εικόνες, μια πρόχειρη παρουσίαση της νομοδότησης, υπογράμμισα τα σημαντικότερα προβλήματα και ελπίζω να έχουμε κάτι τελικά στα χέρια μας που να βελτιώνει την κατάσταση για τις μετανάστριες να τις βοηθήσουμε για την πρόσφαση στην αγορά εργασίας και την κατάσταση επίσης για την κάλυψη την κοινωνική ασφάλιση ίσως μπορούμε να βελτιώσουμε και θα ευχαριστώ πάρα πολύ για τυχόν σχόλια. Ε, κυρία Μορβάη, ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Εισηγήτρια, είναι πάρα πολύ λεπτομερής αυτή η παρουσίαση που ακούσαμε. Η παρέμβασή μου ε, ακολουθεί την πρώτερή μου παρέμβαση. Μιλάμε για τα δικαιώματα των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα ε, υπήρξε ε, θολή εικόνα. Αναφέρθηκε ότι οι γυναίκες, οι μετανάστριες δεν είχαν μεγάλα προβλήματα, δεν υπέφεραν αποστερείς και από φτώχεια σαν να μιλάγαμε όμως για τις γυναίκες που φτάνουν από, από μακρινές χώρες. Πρέπει να δούμε κατά μάτια, στα μάτια αυτά τα προβλήματα και αυτή την τροπή. Στα νέα κράτη-μέλη, μετά την περίοδο του κομμουνισμού, πολλές γυναίκε γυναίκες που μεταναστεύουν στις παλιές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα όσον αφορά τη φτώχεια, στέρηση από δικαιώματα, πολύ χαμηλούς μισθούς, πολύ χαμηλές αμοιβέ και πάνε να εργαστούν σαν babysitters, σαν ε, καθαρίστριες ε, οι συνθήκες είναι πολύ ασαφείς, πολύ συχνά πέφτουν θύματα κυκλωμάτων πορνείας, εμπορίου λευκής αρκός κλπ. Δοθέντως ότι συζητούμε τώρα μία έκθεση όσον αφορά την μετα... τις μετανάστριες, ας μιλήσουμε ξεκάθαρα για αυτό το φαινόμενο που αφορά τις γυναίκες που προέρχονται από τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής και Ευρώπης και πηγαίνουν προς τις παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται περί ε, κοινοτικής μετα... ενδοκοινοτικής μεταναστεύσης και θα πρέπει να δώσουμε την ίδια προσοχή και για αυτές τις μετανάστριες, για αυτές τις γυναίκες. Ποιος θα εγγυηθεί σε αυτές τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και τη διαμονή τους στις χώρες υποδοχής πρέπει να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση και τη γυναίκε από τι τρίτε χώρε και πρέπει να υπάρχει μάλλον με αντιμετώπιση των γυναικών από τα νέα κράτη-μέλη να είναι ίδια με την αντιμετώπιση των γυναικών των χωρών ε, τη ίδια τη χώρα υποδοχή. Λοιπόν, πρέπει όλα αυτά να τα συζητήσουμε. Θα πρέπει να δούμε πώς ζουν οι μετανάστρες, κυρίως οι μετανάστρες που από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες πάνε στις παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να προσθέσω και κάτι. Δεν αρκεί απλώς ένα ερωτηματολόγιο για να δοθούν απαντήσεις. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να ρωτήσουμε ποια δικαιώματα μπορούν να απολαύσουν. Μπορούν να έχουν παιδιά. Όταν έχουν παιδιά, τι δικαιώματα έχουν. Ποια είναι τα δικαιώματα που μπορούν να απολαύσουν αυτέ που μεταναστεύουν και πάνε σε άλλη χώρα για να μην υποφέρουν από και να μην πέφτουν θύματα των κυκλωμάτων τη πορνεία. Να τα συζητήσουμε αυτά. Α πάψουμε να λέμε ψέματα. Να πούμε ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι χώρε προορισμού για τη μετανάστευση και μόνο. Διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποια κράτη-μέλη είναι χώρε προέλευση, καταγωγή για τη μετανάστευση και όχι μόνο χώρε προορισμού. Ευχαριστώ. Α ακούσουμε την κυρία Ζαμπόσκα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Σένιτσιν για τη δουλειά που έκανε και θα ήθελα ε, εξ αρχής ε, σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση να ε, δηλώσω την σύμφωνη γνώμη μου. Ε, μία μικρή παρατήρηση μόνο. Πρέπει να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στην ελεύθερη κυκλοφορία ε, των ατόμων αφενός και των εργαζομένων αφετέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μάλλον των ατόμων και των εργαζομένων αφενός και των μεταναστών αφετέρου. Όταν μιλάμε για άτομα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Η κυρία Σένιτσιν καθιστά σαφές ότι οι μετανάστριες που τηρούν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι νομίμως διαμένοντες μετανάστες, δεν πρόκειται για παράνομη, λαθρέα μετανάστευση. Αυτές οι γυναίκες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα εμπρόθεσμα να καταθέσω και τρεις ε, τροπολογίες. Η κυρία Σέρινσιν ε, μας μιλά για την αναγκαιότητα να ενισχύσουμε στις ε, πολιτικές απασχόλησης και στις κοινωνικές πολιτικές τον ρόλο που προσδίδεται στις γυναίκες. Ενδεχομένω θα έπρεπε να προσθέσουμε το εξή. Η αναγνώριση τη οικογενειακή ζωή για τα συντάξιμα δικαιώματα εν τη αυτή περίπτωση, διότι πολλέ μετανάστρε ασχολούνται με μέλη τη οικογένειά του, με τα παιδιά του για μια συγκεκριμένη περίοδο και εμεί επιμένουμε αυτή η περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κατοχυρώνεται ω συντάξιμο δικαίωμα. Και πιστεύω ότι εφόσον το επιδιώκουμε αυτό για τι γυναίκε Ένωση, θα πρέπει να το επιδιώκουμε και για τι μετανάστριες. Δεύτερον, συμφιλίωση τη οικογένειακή και τη επαγγελματική ζωή, Και εδώ έχουμε πολλά προβλήματα για τις ε, υπηκόους τη Ένωση, ε, και άρα θα πρέπει να επιμείνουμε να ισχύσουν οι ίδιοι ακριβώς κανόνες και για τις μετανάστριες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ας ακούσουμε την κυρία Νικολάη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα. Παρότι είναι λίγο αδύναμη η συνεισφορά του η εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ρεαλιστικό ζήτημα. Δυστυχώς, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε είμαστε αντιμέτωποι με αυτό το ζήτημα υπό δύο ε, μορφές, δύο εκφάνσεις. Έχουμε εσωτερική μεταναστευση από φτωχότερε χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, παραδείγματο χάρη. Πρόκειται για εσωτερική μετανάστευση υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυστυχώς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με υπηκόους των χωρών στις οποίες μεταναστεύουν. Όμως πρέπει να αγωνιστούμε για υιοθέτηση κοινή προσέγγισης παρότι αυτό δεν είναι στα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική πολιτική δηλαδή, παρόλα αυτά πρέπει να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη, να αναγνωρίσουν ε, την ισχύ των ιδίων προτύπων για όλες τις υπηκόσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η άλλη έκφανση του ίδιου ζητήματος είναι οι μετανάστριες από τρίτες χώρες. Ε, το ίδιο θα πρέπει να επιδιώξουμε και για αυτές. Είναι απαραίτητο να γύρουμε και άλλα δύο σημαντικά ζητήματα. Χρειαζόμαστε μία λύση για την ε, παραοικονομία, την, ε, κυρίως ε, για τις γυναίκες τίθεται σημαντικότατα το ζήτημα της πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων. Το, όπως είπε και η κυρία Ζαμπόσκα, η άλλη πτυχή του ζητήματος είναι εσωτερική, δηλαδή οι γυναίκες είναι οι πλέον ευάλωτες στο, ασφαλ... στο συνταξιδοτικό σύστημα. Υπάρχει μεγάλη ανισορροπία. Και θα διενεστεί η κατάσταση αν δεν παρέμβουμε. Αφήστε που είναι επικίνδυνη. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων τους είναι σημαντική γιατί είτε μιλάμε για εσωτερική είτε για εξωτερική ε, μετανάστευση Αυτές οι γυναίκες οικιακές βοηθείως επιτοπλίστων αναγκάζονται να δεχτούν τη δουλειά ακριβώς διότι δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά τους προσόντα. Δεν έχουν και κίνητρο στη συνέχεια για να εργαστούν αποτελεσματικά. Χρειαζόμαστε μια ενημερωτική εκστρατεία για να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους οι γυναίκες, να κατάρτιση για την εφαρμογή της διαδικασίας απάλληψης ε, της διακριτικής μεταχείρισης. Μετά από αυτή τη γνωμοδότηση που είναι εξαιρετικά σημαντική κατά τη γνώμη μου για την Επιτροπή μας. Μπορούμε να ε, εργαστούμε περαιτέρω για αυτό το ζήτημα, ε, γιατί όχι και μια δημόσια ακρόαση για να αναλύσουμε ε, την κατάσταση στα κράτη-μέλη για, την για το θέμα της εσωτερικής μετανάστευσης και να μελετήσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν δηλαδή ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τους συμπεφωνημένους κανόνες, ε, τι συμβαίνει. Πάντως, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση. και η θεώρηση των πραγμάτων που μας προτείνεται μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Μετά και τις τροπολογίες στην εξέταση αυτό νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ χρήσιμη έκθεση. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Αλτάρο, πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Αλτάρο, παρακαλώ, ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και ασχολούμαι με θέματα μετανάστευσης, ε, παράνομης μετανάστευσης και ε, ε, ένταξης. Πρώτα θα αναφερθώ σε πολίτες τρίτων χωρών και μετά περισσότερο στα θέματα του φύλου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να ε, μιλήσουμε για την ένταξη, πολύ συχνά συζητείται αυτό το θέμα σε επίπεδο συμβουλίου με τα κράτη-μέλη, όχι και τόσο συχνά όμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και προσβλέπουμε με ενδιαφέρον ε, στην έκθεσή σας. Το θέμα των υπηκών τρίτων χωρών αφορά τα κράτη-μέλη. Μιλώ για πολίτες τρίτων χωρών πάντα. Και η ένταξή τους γίνεται και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά συνδέεται και με νομοθεσία και πολιτική που ορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο. Ε, και μεταξύ αυτών είναι και η οδηγία για την ε, αμοιβή και ε, για την νόμιμη μετανάστευση. Ας πούμε, η ενιαία άδεια παραμονής ορίζει ενιαία δικαιώματα και ένα πλαίσιο. Αυτά είναι ε, στοιχεία που βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και στην ευημερία. Αυτό ε, επιβεβαιώθηκε και με την νέα βάση, ε, νομική βάση με τη συνθήκη της Αβώνας 79.4 είναι το άρθρο για στενή συνεργασία και θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά την ένταξη, ε, δίνει το πλαίσιο για την παρακολούθηση ε, η Ένωση, για τη συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Και σε επίπεδο διακυβέρνηση ε, μπορεί να δώσει και κίνητρα με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα. Στα πλαίσια αυτά, πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ένταξη ε, και δείχνει και τις προκλήσεις που έχουμε αλλά και το περιθώριο δράσης. Αφορά πάντα τους νόμιμους μετανάστες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία ε, των πολιτών ε, μαθαίνοντας τη γλώσσα, έχοντας πρόσβαση στην εκπαίδευση και θεωρώντας ότι ανήκουν σε αυτή την κοινωνία. Επίσης έχει και συστάσει για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν μαθήματα τη γλώσσα τους, να δίνουν προσοχή ε, και να λαμβάνουν υπόψη και την επαγγελματική ζωή των μεταναστών. Δηλαδή τα μαθήματα να γίνονται σε ώρες που ε, είναι ελαστικές και ευέλικτες. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα προσόντα με ενεργό πολιτική για την εργασία και για την αγορά εργασίας για να συμμετέχουν μετανάστες ή μετανάστριες οι γυναίκες να αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία, να χειραφετούνται και να προοδεύουν. Δικαιώματα λοιπόν των μεταναστών θα πρέπει να τα γνωρίζουν και ε, να γνωρίζουν ταυτόχρονα και τις υποχρεώσεις. Θα πρέπει όμως και οι μετανάστες να δείχνουν προθυμία ένταξη στην κοινωνία που ζουν και σεβόμενοι τις αρχές και τις αξίες της. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ο σεβασμός τους κατοχυρώνονται στη συνθήκη. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ε, μια μάχη κατά των διακρίσεων και να μπορέσουν οι μετανάστες να μάθουν ποιε είναι οι αρχές, οι αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη-μέλη και να ενισχυθούν αυτές οι προσπάθειε. Η ατζέντα αυτή λοιπόν ε, ε, αφορά την ένταξη, αλλά η ένταξη γίνεται σε τοπικό επίπεδο και εκεί πετυχαίνει, αποτυχαίνει. Ε, συνεργασία σε αυτή την περίπτωση με την Επιτροπή Περιφερειών είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης η ατζέντα τονίζει τον τρόπο με τον οποίο, και είναι σημαντικό αυτό, συμμετέχουν οι χώρες προέλευσης ας πούμε, θα πρέπει να τους βοηθούν πριν την αναχώρησή τους ε, με όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, τι ισχύει στη νέα χώρα, τι διατάξεις υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθηση, είπαμε, συγκριτική αξιολόγηση με κοινού δείχτες για να ελέγχονται τα αποτελέσματα της πολιτικής ένταξης των μεταναστών. Η πρόταση είναι να είναι πιο συγκρίσιμα τα στοιχεία στην Ένωση για να μπορούμε να ελέγχουμε τα αποτελέσματα της ένταξης μεταναστών και να υπάρχει και ενίσχυση της κοινοτικής μεθόδου. Τέσσερα είναι τα σημαντικά σημεία, οι τομείς μάλλον, η εργασία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ε, ένταξη και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Ε, ωστόσο οι μετανάστες είναι ακόμα σε δυσχερέστερη θέση ε, σε ό,τι αφορά την κοινωνική συμπερίληψη, την εργασία και την παιδεία σε σχέση με τους γηγενείς. Η ανεργία μεταξύ των μεταναστών είναι 10% ε, περισσότερη από ό,τι μεταξύ των αυτοχθόνων. Και υπάρχουν και άλλοι δείκτες σχετικά με την παιδεία κλπ. Σήμερα οι μετανάστριες κυρίως ε, εργάζονται σε άτυπες επισφαλείς ή προσωρινές μορφές εργασίας, κακοπληρωμένες, ακόμα και όταν είναι πλήρους απασχόλησης. Εργαζόμαστε για να εκπονήσουμε ευρωπαϊκά μοντέλα που θεωρούμε σημεία αναφορά ευέλικτα και μπορούν να υιοθετηθούν και χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη ε, ανάλογα με τις εκάστοτε προκλήσεις για τη μετανάστευση. Μοντέλα κάνουμε λοιπόν ε, σε τρεις τομείς ενεργή συμμετοχή παντού στη κοινωνία των πολιτών, ένταξη των μεταναστών και μαθήματα γλώσσας. Οι επιτροπές μας ε, δύο φορές το χρόνο ε, διοργανώνουν ε, σεμινάρια και το επόμενο θα γίνει την άλλη εβδομάδα, 16 και 17 Οκτωβρίου και θα ασχοληθεί με θέματα συνεισφοράς των μεταναστών στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο σημαντικό μέσο είναι το Ευρωπαϊκό μέσο ένταξης. Ε, αυτή την περίοδο είναι 125 εκατομμύρια από το 7 μέχρι το 13. 80% ε, δαπανάται σε τοπικό επίπεδο κρατόμελών, αλλά 20% σε κοινοτικό. Είναι ένα φιλόδοξο ταμείο και για το επόμενο διάστημα θέλουμε να διατηρηθεί την επόμενη προγραμματική περίοδο λοιπόν των πολιετών προοπτικών για να υπάρχει μεγαλύτερη ένταξη σε τοπικό επίπεδο από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και μη κρατικούς. Το πρόγραμμα ε, Δάφνη, ας πούμε, αφορά τις πιο ευάλωτες ε, ομάδες γυναικών και είναι προτεραιότητα στις προκηρύξεις διαγωνισμών, υποστήριξη των θυμάτων βίας και ε, στην προτεραιότητα αυτή θα ε, έχουμε ιδιαίτερη πρόνοια για κορίτσια, γυναίκες και μετανάστριες που είναι θύματα βίας. Και το δεύτερο είναι η βία κατά των γυναικών γενικότερα και θα χρηματοδοτήσει έργα για ε, συνειδητοποίηση και υλικό που να προλαμβάνει τη βία κατά των γυναικών. I also to e Επίσης, τα δικαιώματα των θυμάτων και η αντίστοιχη οδηγία που εγκρίθηκε το 2010, η οδηγία για την πρόληψη και καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, του τράφικινγκ που εγκρίθηκε το 2011 και επίσης η κρίζωση του τράφικινγκ που ε, πρόσφατα εγκρίθηκε το 2012. Αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα και αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη πενταετία. Το 15% των εργαζομένων που φροντίζουν ηλικιωμένου σήμερα στην Ένωση είναι συχνά μετανάστες και μάλιστα μετανάστριες. Εργάζονται με πολύ βαρύ ωράριο, λίγη ελευθερία και λίγη δυνατότητα να ενταχθούν στην κοινωνία. Και δεν είναι η πρώτη τους επιλογή, αλλά είναι ανάγκη γιατί χρειάζονται χρήματα και χρειάζονται να εξοικονομούν χρήματα και να στέλνουν εμβάσματα. Και συχνά πρόκειται για προσωρινούς μετανάστες που σχεδιάζουν να επιστρέψουν, δεν θέλουν να φέρουν την οικογένειά τους. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες είναι κύριες που ε, στατεύονται λιγότερο γιατί είναι με τον πόδι στη μία χώρα και με το άλλο στην άλλη. Ούτε ασφάλιση έχουν, ούτε κάθονται όλα αυτά τα χρόνια που χρειάζονται για να ε, ε, κατοχυρώσουν συνταξιδοτικά δικαιώματα. Γυρνάνε στη χώρα τους και ε, η οικογένεια τους στέλνει αλλού, γιατί τους θεωρούν αυτόματη ταμιακή μηχανή. Δεν έχουν καμία δυνατότητα να μείνουν για να πάρουν μια μικρή σύνταξη ε, για να τους προστατεύει στα γεράματά τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε την εισηγήτρια για την ε, καταληκτική της παρέμβαση. Κυρία κυρία είναι θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλια. Θα περιμένω τις τροπολογίες σας και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι συμφωνούμε και ότι θέλουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ε, μας μένει μόνο το χρονοδιάγραμμα. 5 Οκτωβρίου, 5 το απόγευμα. Είναι η προθεσμία ε, για την υποβολή τροπολογιών. 6 Νοεμβρίου είναι η ψηφοφορία στην Επιτροπή και δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόμη για την Ολομέλεια. Κλείνει και το σημείο 12 και πάμε στο σημείο 13 συνεδρίαση των συντονιστών. Αυτό θα γίνει το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτό το σημείο. 14 τελευταίο σημείο προσεχή συνεδρίαση 5 Νοεμβρίου 3 με 6,5 και 6 Νοεμβρίου από τις 9 ως τις 12.30 εξυπακούεται στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ και στο επανειδήμα.